Ε, Από την ομάδα των φιλελευθέρων έτοιμα να οριστεί ο κύριος Κλίντς, μέλος της αντιπροσωπείας με Ελβετία, ε, Νορβηγία και μεικτή κοινοβουλευτική για την Ισλανδία και τον ΕΟΧ. Η κυρία Νακτετάλ για την αντιπροσωπεία με την Ινδία, η κυρία Μούλερ αντιπροσωπεία σχέσεων Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία, η κυρία Χίρς στην Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Από την ομάδα EFTT ο πρόεδρος έλαβε αίτημα για διορισμό του κυρίου Μότεν στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων Ελευθεριών και Δικαιοσύνης, στην Επιτροπή Γυναικών και στην Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τη φοροποφυγή, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρατηρήσεις έχετε. Εγκρίνονται λοιπόν οι διορισμοί αυτοί.